Uh, have attention, please, and everybody. We are no longer in vacation time, so let's get started. Καλησπέρα σε όλους. Έχουν τελειώσει οι διακοπές, οπότε ας ξεκινήσουμε. Σημειώνω κάποιες απουσίες. Ε, δεν αιτιολογούνται όλες από την προεκλογική εκστρατεία στη Γερμανία. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. το σημείο 26 για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των ομάδων θα καταργηθεί διότι δεν υπάρχει τίποτα προς αναφορά από την τελευταία συνάντηση υπάρχουν αντιρρήσεις όχι υιοθετείτε να σας ανακοινώσω ότι η συνεδρίαση αυτή θα προβάλλεται ζωντανά μέσω web streaming ε, οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες για όσοι ενδιαφέρονται πρόσφατες ε, ειδήσει για το διεθνές ε, εμπόριο πρώτα απ' όλα ο νέος γενικός διευθυντής Ρομπέρτος Βίντο έκανε την ομιλία του, την πρώτη του ομιλία στο Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και έκανε έκκληση για το συνάντηση στον Παλί οι τελευταίες εξελίξεις για τις πιέσεις της Ρωσίας επί των χωρών της Ανατολικής Ατρικής Σχέσης διαδοθήκαν ε, ειδήσει ότι επιβάλλουν στοχευμένα μέτρα κατά της Λιθουανίας γιατί φυσικά η Λιθουανία κατέχει αυτή τη στιγμή την Προεδρία του Συμβουλίου. Η Επιτροπή με ενημέρωσε ότι οι νομικές διαδικασίες της ε, Συμφωνίας ε, Ελεύθερων Συναλλαγών με τη Σιγκαπούρη έχει ολοκληρωθεί την τελευταία εβδομάδα. Θα, ξεκινήσουμε με την, θα προχωρήσουμε με την προσυπογραφή της ε, συμφωνίας που προγραμματίζεται να λάβει η χώρα στις 20 τρέχοντος στη Σιγκαπούρη. Η μετάφραση έχει ήδη ξεκινήσει σε όλες τις ε, γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδέχεται να ολοκληρωθεί πριν τα τέλη του έτους. Ενώ δεν το περίμενε κανείς. Αυτό θα ανοίξει το δρόμο για την υπογραφή και για την ε, κλήση αυτού του κοινοβουλίου για επικύρωση. Επιταχύνεται λοιπόν η διαδικασία αφού ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις. Επιτυχώς. Σημείο 3. Ο σημερινός ε, τριμερής διαλόγος, ε, κανονισμός ε, που αποτελεί κομμάτι του πακέτου ευθυγράμμισης με το νέο κανονισμό επιτροπολογία και της κατευσίδωτης πράξη όπως ορίζονται από τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Ωστόσο, εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διευρύναμε το εύρο των τροπολογιών με ουσιαστικέ τροπολογίες σε σχέση με στοιχεία, σημεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς παρακολούθηση. Αυτό εγκρίθηκε στο Κοινοβούλιο και δεν είμαστε σε θέση να απορρίψουμε αυτή την τροπολογία. Υπάρχει ισχυρή αντίθεση τόσο από την Επιτροπή όσο και από το Συμβούλιο. Εμείς όμως μένουμε στην εντολή μας. Αναμένουμε να προγραμματιστεί ο επόμενος τριμερής διάλογος. Το ζήτημα αυτό θα είναι περίπλοκο μεταξύ της Επιτροπής και του Συμβουλίου, ωστόσο ήθελα να δηλώσω τόσο στην Επιτροπή όσο και στο Συμβούλιο ότι θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα. Διαφορετικά το πρόβλημα μπορεί να γίνει πολύ χειρότερο για το σημείο 4 δύο αρχεία δεν είμαστε υπεύθυνοι επιτροπή για αυτά είναι η επιτροπή Γιούρη εμείς αποφασίσαμε να συντάξουμε γνωμοδοτήσεις για τη Γιούρη εισηγητής και των δύο είναι ο Τζος διότι αποτελούν ε, πακέτο δέσμη το πρώτο αφορά την προσέξη των νομοθεσιών των κρατομολών όσον αφορά τα εμπορικά σήματα, αναδιατύπωση μιας οδηγίας του 2008 και η δεύτερη αφορά κανονισμό του Συμβουλίου, τροπολογία του, του κανονισμού του Συμβουλίου για το κοινοτικό εμπορικό σήμα. Στενά λένε τα, τα δύο θέματα αυτά. Ε, έχουμε ένα συγκεκριμένο θέμα εδώ, δηλαδή τη μετακόμιση παραποιημένων αγαθών. Κύριε Κουτάς, έχετε το λόγο για να παρουσιάσετε. Εδώ εξετάζουμε τις τροπολογίες. τροπολογίες βρίσκονται στα έγγραφα που έχετε μπροστά σας. Ας συζητήσουμε λοιπόν τις τροπολογίες. Δίνω το λόγο στον Ζωος Κουτάς για να ξεκινήσει η συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπω αναφέρατε, οι προτάσει ε, τη Επιτροπή έχουν στόχο να καταστεί το σύστημα για την καταχώρηση των ευρωπαϊκών σημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιο αποτελεσματικό, αλλά και για να είναι συμπληρωματικά με τα ε, διεθνή συστήματα εμπορικών σημάτων. Στις δύο γνωμοδοτήσεις επικεντρώθηκα αποκλειστικά ε, στις πτυχές που αφορούν ε, το εμπόριο και ε, σε ό,τι αφορά την μετακόμιση των παραποιημένων προϊόντων για την καταπολέμηση της πώλησης τους μέσω του διαδικτύου. Μια πρόταση για την διεύρυνση του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που κατέθεσαν τροπολογίες για αυτές τις διαγνωμοδοτήσεις. Ιδίω χάρηκα που είδα τροπολογίε για την προστασία ε, της πρόσβασης ε, στα γενώσιμα φάρμακα και θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Επίσης, αποφάσισα να τροποποιήσω ελαφρώ το σχέδιο γνωμοδότηση για να αντικατοπτρίζεται και ο προβληματισμό ότι η ε, παροχή προϊόντων σε διαμετακόμιση ίσως να μην συνάδει με τους κανόνες του ΠΟΕ. Έτσι είδα ότι η ε, γνωμοδότρια της Τζούρι, η Σεσίλια Βίξτρομ, άλλαξε τη θέση της για να πει ότι θα πρέπει να δίδονται αποδείξεις του εμπορικού σήματος και της εγκυρότητάς του στο, στην χώρα προορισμού. Αυτό θα πρέπει να εξακολουθήσει να συζητείται, θεωρώ, ως θέμα. Όπως είδα και η Αμάλια έχει καταθέσει τροπολογία για αυτό το τμήμα του κειμένου. Μένω ανοιχτός ε, σε συζήτηση να δούμε ποιο είναι ο κατάλληλο συμβιβασμός. Όμως, όπως σας έχω πει, νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε ακριβώς στι πτυχέ που αφορούν το εμπόριο και να μην επεκταθούμε περαιτέρω. Γιατί αυτή είναι η αρμοδιότητα της Επιτροπής μα. Ευχαριστώ. Ναι, βεβαίω, έχετε δίκιο, ο Αυτή η γνωμοδότηση αφορά τα ζητήματα επί του εμπορίου. Να δώσουμε το λόγο στους ασκιόδης. ΕΛΚ, όχι. ΑΛΔΕ, όχι. Όχι μεταρρυθμιστές. Αμαλία, από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις προσπαθειές του και ελπίζω να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Εμείς γενικά στερίζουμε την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο εισηγητής, ωστόσο θεωρούμε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη φιλοδοξία από την Επιτροπή μας για να, υπάρχει πιο, ε, να υπάρχουν πιο δίκαιοι και ισότιμοι αλλά και κατανοητοί κανόνες. Πρέπει να αλλάξουν κάποιες από τις συντολογικές σκέψεις στα άρθρα για να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια και εύρυθμη λειτουργία του εμπορίου. Πρώτα έχουμε τη διαδικασία της διματακόμισης. Αρχικά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αποφασίσει, αποφανθεί επί των κατασχέσεων και έχει θεωρήσει ότι είναι παράνομες και θα πρέπει να προστατεύουμε τους Ευρωπαίους καταναλωτές και όχι μόνο τους, και όχι τους καταναλωτές που δεν είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνοι οι πολίτες λοιπόν που δεν είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βασίζονται στις δικές τους, ε, στα δικά τους ε, νομικά συστήματα. Εμείς δεν μπορούμε λοιπόν να δαπανούμε πόρους για εκείνους. Δεν θεωρούμε ότι είναι κατάλληλο να λέμε στο 19 τα συγκεκριμένα προβλήματα ε, στα εμπορικά σήματα και στο διαδίκτυο. Είναι μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη διαδικασία και ως Ένωση θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να επιληθούν τα υφιστάμενα νομικά ζητήματα. Είναι ένα γνωστό ε, πρόβλημα ότι ε, συνεχίζονται αυτές οι διαδικασίες και υπάρχουν πάρα πολλές ε, υποθέσεις στις εισαγωγές, εξαγωγές και ούτω καθεξής δεν ε, βοηθά ούτε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, το δίκαιο επί των εμπορικών σημάτων να γίνει ιδιαίτερα περίπλοκο και έτσι μεταρρυθμίσει σε αυτό το δίκαιο δεν ε, είναι η κατάλληλη λύση αυτή τη στιγμή. Το καλύτερο θα ήταν και για τις εμπορικές μας σχέσεις να βασιστούμε σε απλούς κανόνες που να επιλύουν και όχι να δημιουργούν νέες αντιδικίες. εάν υπάρξει ένα μέτρο ε, στα σύνορα, τότε αυτό το πρόσωπο θα φέρει ευθύνη ε, όταν ε, η παρέμβαση αυτή είναι παράτυπη. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Είναι δύσκολο και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αμυνθούν να περισσούν τον αυτό τους απέναντι ακόμα και σε άδικες τέτοιες παρεμβάσεις. Ελπίζω συνάδελφοι να συμφωνήσουν με αυτές τις παρατηρήσεις και να εργαστούμε όλοι από κοινού από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Thank uh, Ευχαριστούμε πολύ από τον Κούα, Χέρμαν Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Ήδη στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων για αυτό το χαρτοφυλάκιο είχαμε συμφωνήσει και είχαμε πει ότι με την προσέγγιση αυτή την οποία ανέπτυξε στοχεύει στην σωστή κατεύθυνση. Και εγώ σε σχέση με τροπολογία μου και πάλι επικεντρώνομαι στο θέμα της διάθεσης των γενώσιμων προϊόντων ώστε να έχουμε σαφής και δεσμευτικά από νομικής πλευράς ε, δυνατότητα δεσμευτική νομικής ασφάλειας που θα δημιουργείται. Αυτά τα οποία έχουμε στη συζήτηση σήμερα είναι επενέσιμα ως προσπάθεια και το βρίσκω και σωστό στην ε, τροπολογία αυτή που έχουμε από τον συνάδελφο να αναφερόμαστε στον ΠΟΕ Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και στον γύρο της ΔΟΧΑ. μπορούμε να συμφωνήσουμε επ' αυτού τότε κερδίζει από πλευράς ποιότητας η έκθεση και έτσι η έκθεση συνολικά μπορεί να αναβαθμιστεί και να συνεισφέρει στην ρύθμιση της αγοράς και να συνεισφέρει σημαντικά. Ευχαριστώ. Time to listen to the... Έχει έρθει να ακούσουμε την Κομισιόν Μάικλ Κάνιχ που βρίσκεστε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλα τα μέλη για την πολύ επικοδομητική συζήτηση και τη συμβολή τους και εμείς φυσικά ανυπομονούμε να συμβάλλουμε περισσότερο με την εργασία μας σε αυτό το αρχείο. Θα ήθελα απλά να αναφέρω δύο σημεία εντάχει το πρώτο απλά για να υπενθυμίσω τη φιλοσοφία μας ε, που, στην οποία στηρίζεται αυτή η πρόταση για τα παραποιημένα αγαθά και τη διαμετακομισή τους. Στόχος εδώ είναι να στείλουμε ένα καθαρό μήνυμα ότι αυτή η μάχη κατά της παραποίησης ε, λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφενός θέλουμε να στοχεύσουμε, να προστατεύσουμε ουσιαστικά τους καταναλωτές εντός της Ένωσης αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο σημαντικό σκέλος. Το να αποφύγουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει κεντρικό σημαντικό κόμβο για τη διαμετακόμιση τέτοιων παραπημένων αγαθών σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο η πρότασή μας είναι πράγματι φιλόδοξη. Προσπαθεί να συμπεριλάβει και τα δύο στοιχεία. Δεύτερον, θα ήθελα να σε επιβεβαιώσω και να υποστηρίξω οποιασδήποτε προτάσεις ε, με τις οποίες θα διευκρινίζεται ότι οι προτάσεις μας, όλες οι προτάσεις μας δεν πρόκειται να επηρεάσουν κατά κανένα τρόπο το εμπόριο γενώσιμων ε, φαρμάκων ή γενικών αγαθών. Ε, πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό προϊόν και συνεπώς εντελώς διαφορετικό ζήτημα, διότι πρέπει να κάνουμε πολύ προσεκτικά μια διάκριση μεταξύ αφενός των γενώσιμων φαρμάκων φάρμακα δηλαδή τα οποία αναπαράγονται με το ίδιο περιεχόμενο, με τα ίδια συστατικά και που θέλουν να, διακρι... να διακρίνονται από το γνήσιο προϊόν, συνήθω με υπό ένα άλλο όνομα, μάρκας και οποιασδήποτε διενέξεις σε αυτό το τομέα αφορούν ουσιαστικά παραβιάσεις διπλωμάτων ευρυστιχνίας. Εδώ μιλάμε για εμπορικά σήματα όμως. Συνεπώς ε, οποιασδήποτε διαφωνίες, διαφορές σε σχέση με γενώσιμα φάρμακα δεν επηρεάζονται από αυτό εδώ το κείμενο. Ωστόσο, αν μιλάμε για παραποιημένα φάρμακα, δηλαδή φάρμακα τα οποία ε, παράγονται παράνομα και των οποίων η προέλευση δεν είναι σαφής, σε αυτή την περίπτωση πιστεύω είναι σημαντικό να προστατεύσουμε τους καταναλωτές από τέτοιου προϊόντα όπου, που διακυβεύουν την ασφαλεία τους. Ό,τι προτάσει έχετε ώστε να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε ότι τα γενώσιμα φάρμακα και το εμπόριο του δεν θα επηρεαστούν, ε, θα ήταν ευπρόσδεκτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ζωής Κούτας, ε, περαιτέρω παρατηρήσεις, ναι. Ευχαριστώ ξανά όλους τους συναδέλφους για την συμμετοχή τους. Όπως αντιλαμβάνομαι έχουμε τους ίδιους στόχους. Ας δούμε ε, κατά πώς θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια σωστή διατύπωση ώστε να μείνουν όλοι ικανοποιημένοι. Προτείνω την επόμενη εβδομάδα να ζητήσουμε να λάβει χώρα μια συνάντηση και με την Κομισιόν για να δούμε κατά πόσο θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε όλοι. Ευχαριστώ και πάλι. Επόμενο βήμα της διαδικασίας ψηφοφορία των τροπολογιών στην Επιτροπή στις 14 Οκτωβρίου στην τακτική μας συνάντηση του επόμενου μήνα. Σημείο 6. Μακροοικονομική βοήθεια στο Χασιμητικό Βασίλειο της Ορδανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την οποία είμαι εγώ εισηγητής δεδομένη της κατάστασης σήμερα το αρχείο αυτό θα πρέπει να αποφασιστεί γρήγορα. Έχετε το σχέδιο έκθεσης ε, μπροστά σας, όπως γνωρίζετε όλα τα μακροοικονομικά ζητήματα διευκολύνθηκαν ιδιαίτερα μετά από τη συμφωνία μας με το Συμβούλιο επί ενός ε, πλησίου που υιοθετήθηκε μαζί με την αποφασή μας για την ε, Ιορδανία. Τώρα λοιπόν το μόνο που μένει είναι να προσαρμόσουμε το πλαίσιο κατά περίπτωση. Έτσι λοιπόν όλες μου οι τροπολογίες αποσκοπούν στην ευθυγράμμιση αυτού του αρχείου που είναι νομοθετικό με το πλαίσιο που, έχει που έχουμε συνεννοηθεί με το Συμβούλιο. σε αυτή την περίπτωση θα ισχύσει η διαδικασία εξέτασης για την υιοθέτηση του μνημονίου κατανόησης διότι μιλάμε για ποσά άνω των 90 εκατομμύριων ευρώ ένα κατόφλιο ουσιαστικά που έχει οριστεί σε αυτό το κοινό μνημονίο με το Συμβούλιο. Συνεπώς ε, λογικά δεν θα υπάρξει κάποια μεγάλη δυσκολία εδώ. Νομίζω ότι γενικά συμφωνούμε με την Κομισιόν ότι αυτή η μακροοικονομική αρρωγή θα πρέπει να παρασκευθεί στην Ιορδανία. Αυτή είναι λοιπόν η πρότασή μου. Ας ανοίξουμε λοιπόν τώρα το... συζήτηση. Βλέπω μόνο τον κύριο Πόμερφη, τον Γκουε, τον κύριο Πολ Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σίγουρα συμφωνούμε. Πιστεύω ότι οι Ορδανοί θα έπρεπε να τύχουν αρρωγή. Το θέμα είναι πώς θα τους βοηθήσουμε, υποθέτω. Συμφωνώ σε σχέση με τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Να τονίσουμε το θέμα της δημοκρατίας, ε, της ε, ένομης τάξης δικαίου, του κράτους ε, δικαίου. Αλλά έχουμε και ένα θέμα θεμελιώδες εδώ για το πώς θα πρέπει να δοθεί αυτή η βοήθεια και το μνημόνιο συνεννόησης ε, παράλληλα με τα προγράμματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το αν αυτή η χρηματοδότηση θα προβλέπει και αναδιάρθρωση της οικονομίας με ένα νεοφιλελεύθερο τρόπο ή όχι και αν αυτό ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Ιορδανών ή όχι. Διότι πριν από ένα χρόνο και λιγότερο από ε, πριν από ένα χρόνο περικόπηκαν οι επιδοτήσεις, οι ενισχύσεις σε σχέση με την Ιορδανία. Ο λόγος ήταν ότι αυξήθηκαν οι τιμές των καυσίμων πάνω από 50%. Τεράστιες διαδηλώσεις ε, έγιναν, υπήρξαν νεκροί και άλλα μέτρα παρόμοια <clears throat> μια και υπάρχουν χώρες όπως και η Ιορδανία που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και βλέπουμε το καρότο το χρησιμοποιούν αλλά και το μαστίγιο επίσης και βλέπουμε εδώ το μνημόνιο ε, συνεννόησης ε, με ένα νεοφιλελεύθερο πνεύμα που σίγουρα αφορά και τους στόχους εκείνους ε, που όταν ξεκίνησαν οι, τα κινήματα, οι επαναστάσεις αυτές, που σίγουρα πρέπει να πούμε ότι συνδέονται με τα δημοκρατικά δικαιώματα, με τα θέματα ευημερία, αλλά πρέπει να δούμε και τις ε, επιπτώσεις ε, που ε, συνεπάγονται οι μεταρρυθμίσεις αυτές που επιβάλλονται στην Ιορδανία. Πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί λοιπόν και να δούμε όλες αυτές τις πτυχές και τις επιπτώσεις τους. Πρόεδρος, δεν ζητεί άλλος να παρέμβει. Ας ακούσουμε τώρα την Επιτροπή. Κρίστοφ Βάγνερ, παρακαλώ. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης και για την έκθεση που ε, ευθυγραμμίζεται και με την ε, δήλωση των συνομοθετών. Επί της ουσίας συμφωνούμε απόλυτα με την έκθεση. Έχουμε κάπως, ε, κάποια ελάσσονος σημασίας σχόλια ή τροπολογίες που γραπτά θα σας τα διαβιβάσουμε στη γραμματεία σας όπως αναφέρθηκε για την Ιορδανία είναι πάρα πολύ σημαντικό να δοθεί αυτή η βοήθεια, η αρρωγή τάχιστα πολύ γοργά. Η σύγκρουση στη Συρία έχει προκαλέσει 600.000 ε, ε, πρόσφυγες και αυξάνονται. Επίσης η ροή φυσικού αερίου από την Αίγυπτο εξακολουθεί να ε, βρίσκεται υποδιακοπή, έχει διακοπή και δεν πρόκειται να επανέλθει σύντομα. Γι' αυτό λοιπόν έχει πολύ αυξημένε τιμέ καυσίμων η Ορδανία σε σχέση με άλλε χώρες. Και αυτό έχει οδηγήσει σε ε, οξύτατα προβλήματα όσον αφορά ελλείμματα κτλ. Η κατάσταση είναι λοιπόν κατεπίγουσα και πρέπει να τύχει βοήθειας. Και όσον αφορά τους όρους, οι όροι και οι προϋποθέσεις θα αφορούν θέματα διαχείρισης και δημόσιας χρηματοδότησης. Και Είχαμε <clears throat> προηγούμενες συζητήσεις παραγωγικές ε, με τις, ε, τους κυβερνητικούς εκπροσώπους. Δεν φαίνεται να υπάρχουν επίμαχα θέματα για τα θέματα αρρωγής. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιου. Δεν υπάρχουν προβλήματα ή τριβές σχετικά. Θα είναι λοιπόν σημαντικό να μπορέσουν αυτές οι συζητήσεις να γίνουν μέχρι τα τέλη του έτους ή δυνατόν. Γνωρίζω ότι η μερίσια διάταξη και οι διαδικασίες ε, Ήδη ακολουθούνται επιταχυμένες ε, γοργές διαδικασίες για πράγμα για το οποίο είμαστε ευγνώμονες. Αν καθυστερούσαμε θα ήταν πολύ δύσκολο να ληφθούν οι αποφάσεις αυτές εφέτος ακόμα θα σας απευθύναμε έκκληση παρότι έχει επιταχυθεί η διαδικασία αν θα μπορούσατε μετά τον τριμερή διάλογο κατά τα τέλη Οκτωβρίου να περάσει το θέμα προσέγγισης έγκριση στην Ολομέλεια στη Σύνοδο του Οκτωβρίου. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή την έκθεση και δεσμευόμαστε από πλευρά τη Επιτροπής να προχωρήσουμε σε σχέση με αυτό το θέμα όσο το δυνατόν ταχύτερα. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι κάναμε κάθε προσπάθεια, κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας με τον καλύτερο τρόπο για να προχωρήσει αυτό το χαρτοφυλάκιο. Και για τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το ότι αυτή η αρρωγή κατεπηγόντως χρειάζεται στην Ιορδανία και αν θα μπορούσε το Κοινοβούλιο να κάνει ό,τι περνά από το χέρι του να επιταχύνει γοργά. Λαμβάνεται υπόψη λοιπόν, για να λάβουμε υπόψη αυτά θα προσαρμοστούμε σε, αυτή, σε αυτό το αίτημα. Και τον Οκτώβριο λοιπόν, 14 Οκτωβρίου, θα έχουμε την τακτική μας συνεδρίαση ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή και θα προσπαθήσουμε και πάλι για άλλη μία φορά να κάνουμε αυτή την προσπάθεια να εγγραφεί το θέμα στην ημερήσια διάταξη της περίοδου συνόδου το δυνατόν ταχύτερα. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 24 Σεπτεμβρίου 18.00. 6 το απόγευμα. Τώρα, θέματα 7 και 7α όσον αφορά τα χαρτοφυλάκια που έχουμε πάλι το ίδιο θέμα ενώπιόν μας. Απόφαση Συμβουλίου σχετικά και τροποποίηση του κανονισμού και τα δύο αφορούν την αποκαλούμενη διαδικασία Kimberley όσον αφορά την ε, πιστοποίηση και την ε, εμπορία των ακατέργαστων διαμαντιών. Μίζων πρόοδος όσον αφορά αυτό το θέμα, δηλαδή με άλλα λόγια χρήση των ε, αδαμάντων για να, χρησιμο... να χρηματοδοτούνται κάποιες σειράξεις αγορά όπλων κτλ. Η Γρινλανδία, ε, μια και ε, σε σχέση με την ε, επικράτειά τους δεν είναι ανεξάρτητη χώρα, δεν είναι κυρίαρχο κράτος και έτσι δεν μπορούν να είναι μέρος της συμφωνίας και βλέπουμε ότι η εφάνταστη προσέγγιση των, της νομικής υπηρεσίας και του Συμβουλίου και της Επιτροπής, οι νομικές μας υπηρεσίες με άλλα λόγια τι έκαναν. Σχεδίασαν μια δυνατότητα να επιληθεί αυτό το πρόβλημα ώστε η Γρυλανδία να μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στην ε, Ένωση. Η Γρυλανδία που δεν είναι κυρίαρχο κράτος εγώ είμαι ο εισηγητή ε, για αυτό το θέμα. Είμαστε η αρμόδια επί τη ουσία ε, κοινοβουλευτική επιτροπή. Απόλυτα υποστηρίζω αυτή την πρωτοβουλία και ή δυνατόν πιστεύω ότι θα έπρεπε όλες οι χώρες και οι επικράτειες ε, και τα διαμερίσματα που σε σχέση με τα διαμάντια θα πρέπει να υπάγονται στις διαδικασίες του σχεδίου πιστοποίησης Κίμπερλι, ώστε να μπορεί να διασφαλίζεται ότι θα έρχονται από αξιόπιστες πηγές ε, χωρίς οποιαδήποτε κατάχρηση. Και σε σχέση λοιπόν με αυτό το θέμα της ε, Γρυλανδίας θα πρέπει να, να δώσουμε την υποστήριξή μας, αξίζει να υποστηρίξουμε το αίτημά της και γι' αυτό ακριβώς η πρότασή μου να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ώστε να δοθεί μια θετική λύση, να διευθετηθεί με θετικό τρόπο αυτό το ζήτημα, αυτό το αίτημα της Γρυλανδίας. Επίσης ε, είναι η ευκαιρία αυτή ώστε το Κοινοβούλιο να ενταχθεί, να υπαχθεί σε αυτή την πολύ σημαντική διαδικασία λαμβάνοντας υπόψη τις ευθύνες και την ευθύνη που θα έχουμε μετά την συνθήκη της Λισαβόνας που ισχύει πλέον. Εν πάση περιπτώσει δεν θα μπορούσα να απόσχω από το να συμμεριστώ μαζί σας κάποιες ανησυχίες και επιφυλάξεις όσον αφορά γενικότερα την κατάσταση της διαδικασίας σε Κίμπερλι. Άκουσα ότι υπάρχει μια, ένας συνασπισμός που βρίσκεται επικεφαλής. Δεν θα ήταν δυνατόν να αφήσουμε λοιπόν, πιστεύω, αυτό το σύστημα και τη μέθοδο ιχνηλασιμότητας ανείχνευσης ε, να μην λειτουργήσει όσον αφορά τους ε, ακατέργαστους αδάμαντες. Το αντίθετο θα έπρεπε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύσουμε αυτό το καθεστώς ε, ανείχνευσης και ιχνηλασιμότητας. Και με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να πούμε ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία αυτή, ώστε να εισακουστεί η φωνή του Ευρωκοινοβουλίου στο πλαίσιο αυτών των δράσεων. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσουμε και την, την Επιτροπή, αλλά δεν έχω όνομα εδώ σημειώσει. Ποιος θα λάβει τον λόγο εξ ονόματος της Επιτροπής παρακαλώ. Ναι, καλώς ήρθατε. Εσείς έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ που παρευρίσκεστε και για την ανταλλαγή απόψεων μαζί μας. Από την Επιτροπή λοιπόν, εσείς. Mr. Herenzo. Ο κύριος Χέρενς ή ο κύριος Κόντας. Correct. Σωστά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συναδελφός μου η Μαριανά Κοντάς και εγώ εκπροσωπούμε την Υπηρεσία Εξωτερικής Πολιτικής της Κομισιόν και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε εσάς καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής ε, Διεθνούς Εμπορίου που δίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ευκαιρία να παρουσιάζει τις προτάσεις της από σήμερα. Πριν μπούμε στις λεπτομέρειες της πρότασης μας. Θα ήθελα να σας δώσω μια σύντομη εικόνα της πιστοποίησης Κίμπερλι. Ε, Και είναι δηλαδή μια εθελοντική κρατική πρωτοβουλία ουσιαστικά για την αναχέτηση του εμπορίου των διαμαδιών που τροφοδοτούν οικονομικά τις ε, παγκόσμιες διενέξεις. Οι διαδικασίες αυτές, Κίμπερλι, αφορούν αυτή την παράνομη διακίνηση αδαμάντων και εξασφαλίζεται με μια διαδικασία πιστοποίησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενιαίος συμμετέχων στο σύστημα αυτό συμμετέχει ως ένα μέλος με όλα τα 27 μέτρα εκπροσωπείται από χώρες ε, όπως το Βέλγιο, έξι χώρες, ε, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Τσεχική Δημοκρατία, Βουλγαρία, Ρουμανία. Οποιαδήποτε αποστολή ακατρέας των διαμαντιών που εισάγεται ή εξάγεται σε και προς οποιοδήποτε κράτος μέλος αποστέλλεται στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επαλήθευση και μόνο στη συνέχεια αποστέλλεται στον τελικό παραλήπτη και επιτρέπει ελεύθερη κυκλοφορία του εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις εξαγωγές. Μια από αυτές τις αρχές ε, εκδίδει ένα πιστοποιητικό Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον το εμπόρευμα πληρεί όλες τις απαιτήσει. του κανονισμού 2368 του 2002. Οι απαιτήσει έχουν ω εξή. Πρώτα απ' όλα τα κατάργαστα διαμάντια πρέπει να έχουν εισαχθεί προηγουμένω νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεύτερον θα πρέπει να βρίσκονται σε περιέκτη που τα προστατεύει από τις εξωτερικές συνθήκες. Το 99% των ε, διαμαντιών του κόσμου παράγονται από συμμετέχοντες στη διαδικασία Κίμπερλι. Αποτελεί λοιπόν σημαντικό παράγοντα για κάθε χώρα που παράγει διαμάντια να συμμετέχει στη διαδικασία του Κίμπερλι. Διαφορετικά δεν τη συμφέρει να εξάγει διαμάντια. Η Γρυλανδία λοιπόν δεν είναι ανεξάρτητη χώρα, συνεπώς δεν μπορεί να συμμετάσχει ως τέτοια στη διαδικασία Κίμπερλι. Να σας πω δύο λόγια για τη Γρυλανδία. Αυτή τη στιγμή 88% του ΑΕΠ της Γρυλανδίας προέρχεται από την αλληλεία και 0,8% μόλις από Ωστόσο, ο αληθικός τομέας της Γρυλανδίας λόγω των περιορισμένων ποσοστώσεων αποθεμάτων και λόγω της κλιματικής αλλαγής γίνεται όλο και λιγότερο αξιόπιστος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι η Γρυλανδία θα χρειαστεί να διαφοροποιήσει την οικονομία της και να δει πώς ε, θα μπορέσει να την αναπτύξει αλλού. Μετά το 2011 η Γρυλανδία κατάφερε να υλοποιήσει ολοκληρωμένη νομοθεσία ώστε να διασφαλίσει ότι οι κάτοικοι της Γρυλανδίας θα υποφεληθούν από τα έσοδα που προερχόνται από τα διάφορα μέταλλα αυτά, μεταφέρονται σε δημόσια ταμεία που είναι απαραίτητα για την οικοδόμηση της απαραίτητης ε, υποδομής. Η παραγωγή διαμαδιών ε, αντιμετωπίζεται πολύ θετικά από την κυβέρνηση διότι προκαλεί ελάχιστες περιβαλλοντικές ζημιές από τα άλλα ορεκτά Ωστόσο, επειδή δεν μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό Κίμπερλι για την εξαγωγή των διαμαντιών της, ε, η Γρελανδία δεν μπορεί να προσελκύσει πιθανού επενδυτές. Στον τομέα εξόρεξη και η δική της πόρη δεν είναι επαρκής για να μπορέσει να ξεκινήσει ορίξεις συμφέρουσες οικονομικά. Να δώσω τώρα το λόγο στην συνάδελφο Μαριάννα Κόνα για να σα εξηγήσει την πρώτη λεπτομερέστερα. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Θα ήθελα να πω δύο λόγια ακόμα για αυτή την ε, ιδιαίτερα εφάνταστη λύση όπως ανέφερε και ο εισηγητής. Η Γρυλανδία, εφόσον είναι και ε, υπερπόντια επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά πόσο θα τη βοηθήσει αυτό να κάνει χρήση δηλαδή, του συστήματος ε, διαπίστευση. Αυτό σίγουρα θα προωθούσε την οικονομική ανάπτυξη της Ιρλανδίας, που είναι και στόχος υπό τις συνθήκες. Σε ό,τι αφορά τι συγκεκριμένες προτάσεις, προτείνονται δύο νομικές πράξεις. Υπάρχει πρόταση για μία νέα απόφαση του Συμβουλίου βάσει του άρθρου 203 για, τη συνθήκη, για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσπίζει ένα συγκεκριμένο καθεστώς για την μετακίνηση ακατάργαστων γεματιών μεταξύ Ιρλανδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει συγκεκριμένα ότι οποιαδήποτε εμπόριο τέτοιων ε, διαμαντιών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιρλανδίας θα πρέπει πρώτα να έχει εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν μεταβεί σε μία από τις έξι αυτές χώρες που αναφέρει ο συνάδελφος. Επιπλέον, ε, μια πρόκληση ήταν επίσης να λύσουμε το πρόβλημα ότι δεν βρίσκεται ε, στο, στην Τελωνική Ένωση όπω ε, άλλε ευρυπώντε περιοχέ και έτσι έπρεπε να βρεθεί λύση για αυτό το ζήτημα. Και μια αξιόπιστη λύση μάλιστα, Ούτω ώστε ε, τα τελωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να δεχθούν ε, του αδάπαντες που έχουν εξοριχθεί ή εισαχθεί στη Γελλανδία βάσει εξαίρεσης και απαλλαγή από την υποχρέωση παρουσίαση ενό πιστοποιητικού KP, κάτι που δεν μπορεί να κάνει με τη χρήση λοιπόν ενός άλλου ε, εγγράφου που αναφέρεται στην απόφαση του Συμβουλίου και περιγράφεται στα παραρτήματα. Αυτό λοιπόν το έντυπο θα χορηγείται από τις ε, αρχές της Γρυλανδίας και θα ελέγχεται από τις ε, Ευρωπαϊκές Τελωνιακές Αρχές κατά την είσοδο και έξοδο. Υπάρχουν και περαιτέρω προϋποθέσεις στην απόφαση του Συμβουλίου ούτως ώστε να αποτελέσει μια αξιόπιστη ε, διαβίβαση των διαμαντιών. Ε, αντικατοπτρίζονται εκεί και όλες ε, οι προϋποθέσεις του κανονισμού. Έχουμε την προπόθεση ότι δεν πρέπει να έχει σπάσει σφραγίδα, για παράδειγμα, ή η η να μα δίνει τα στατιστικά στοιχεία και ούτω καθεξής. Αυτά σε γενικές γραμμές ό,τι αφορά την απόφαση του Συμβουλίου. Εκ παραλλήλου υπάρχουν και κάποιες ε, τροποποιήσεις ε, που απαιτούνται για τον 2068 2002 Το πιο σημαντικό, πιο σημαντική αλλαγή, όπως ανέφερε και ο αξιότιμος εισηγητής, είναι ότι η επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Γρυλανδία θα θεωρούνται η ίδια και αυτή η ε, υπόσταση χωρίς εσωτερικά ε, σύνορα, αποκλειστικά και μόνο για το σύστημα πιστοποίησης. Αυτό είναι και ο πυρήνας ε, της τροποποίησης, μαζί και με κάποιες ίσονος σημασίας αλλαγές σε άλλα άρθρα, όπου προσθέτονται κάποιες, προσθέτονται κάποιες αναφορές στη Γρυλανδία όπου αυτό είναι απαραίτητο και σε κάποιες ε, περιπτώσεις που αφορούν μόνο την εξόριξη διαμαντιών στη Γρυλανδία, που έτσι δεν έχουν εξαρθεί εξ αρχής ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένω δεν μπορούμε να απαιτούμε και την ε, νόμιμη εισαγωγή τους. Δεν μπορεί να αποδεχθεί αλλιώς. Αυτό λοιπόν αφορά μόνο τα διαμάντια που έχουν εξοριχθεί στη Γρυλανδία. Τώρα, δεδομένης της ε, κρισιμότητας ε, και του επίγοντος της κατάστασης, η Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει μόνο αυτέ τις πολύ στοχευμένες αλλαγές. Ε, οι παλιές αναφορές προ Λισαβόνα στην διαδικασία επιτροπολογίας μας οδηγούν στο να πρέπει να έχουμε μια ενοποιημένη κατάσταση. Γιατί και οι συνθήκες προβλέπουν την αυτόματη ευθυγράμμιση των υφιστάμενων εγγράφων. Τούτου λεχθέντος, η Επιτροπή μπορεί να δεσμευθεί ότι θα έχει μια τέτοια ενοποιημένη ε, παρουσίαση του ζητήματος. Ωστόσο, προς το παρόν, εφόσον πρόκειται για ένα επίγον ζήτημα, όπως ανέφερε και η Γερλανδία, θα θέλαμε να μας βοηθήσουν τα αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου να επιλύσουμε αυτό το πρακτικό ζήτημα και πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας. Θα θέλαμε λοιπόν και τη δική σας ε, συνδρομή. Για να απαντήσω εν συντομία στα όσα ανέφερε ο εισηγητή ε, πριν από την παρουσίασή μα, η Επιτροπή αναγνωρίζει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα ε, του Ευρωπαϊκού Εμπορίου και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχετε τις απαραίτητες ε, πληροφορίες για να λάβετε τις αποφάσεις σας. Υπάρχουν πολλές ε, υποχρεώσεις απέναντι στην Επιτροπή για την ε, παροχή πληροφοριών μέσω της διαδικασίας επιτροπολογίας. Είναι και δικαίωμα των νομοθετών αυτό βεβαίως. Στο πλαίσιο που περιγράφεται από αυτά το έγγραφο, βεβαίω και η υπηρεσία μου είναι τεθειμένη να εξετάσει πώ μπορούμε να ενημερώνουμε καλύτερα στο μέλλον το Κοινοβούλιο. Συμπερασματικά, να σα ευχαριστήσω για την προσοχή σα και βεβαίω να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερωτήματα ενδεχομένω έχετε ε, για την διαδικασία Κίμπερλι. Βεβαίω, έχουμε σημειώσει τα ερωτήματα ε, του εισηγητή. Θα θέλαμε όμω να απαντήσουμε μετά τις παρεμβάσεις των υπόλοιπων μελών. Ευχαριστώ. Let's Ας αρχίσει η συζήτηση. Ενδιαφέρονται κάποιοι να συμμετάσχουν σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψε. Ποιοι ζητούν να παρέμβουν. Παρακαλώ, εσείς ευχαριστώ πρόεδρε. Ως κοιόδης εισηγητής για αυτό το χαρτοφυλάκιο συμφωνώ φυσικά με την προσέγγισή σας επ' αυτού και υποστηρίζω. Θα έπρεπε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μπορέσουμε ταχύτατα να δράσουμε μέσα σε ένα χρονοπλαίσιο αποτελεσματικά. Να υπάρξει μια διαφανής ρύθμιση, σαφής και διαφανής ρύθμιση για όλους σε σχέση με το εμπόριο αδαμάντων. Το μόνο ερώτημα που θέλω να διατυπώσω, αλλά δεν, είναι, δεν συνδέεται με αυτό το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, αλλά γενικότερα σε σχέση με το θέμα Κίμπερλι, είναι μήπως θα έπρεπε να δώσουμε κάποια δικαιολογία, κάποια επιχειρήματα από τον εθελοντικό χαρακτήρα σε δεσμευτικές προτάσεις ε, και δεσμευτικού χαρακτήρα ρυθμίσεις που θα έπρεπε με αυτόν τον τρόπο να ε, εντάσσονται σε αυτό το δεσμευτικό πλαίσιο όσοι θα συμμετέχουν. Ευχαριστώ. Freiwilligkeit, εθελοντικός χαρακτήρας, εθελούσια ένταξη σε αυτό το σύστημα, σε αυτό το εγχείρημα. Θεωρούμε ότι είναι θεμελιώδες ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτού του είδους ε, η βάση για αυτή τη συμφωνία ώστε να μπορέσει να σημειωθεί πρόοδος. Τώρα, για κάποιους ε, περιορισμούς ή περιοριστικές ε, διατάξεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη, ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Άλλοι θέλουν να παρέμβουν, όχι. Ευχαριστώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τοποθέτησή της. Έχετε και πάλι τον λόγο αν επιθυμείτε να παρέμβετε για μια πρόσθετη παρέμβαση από πλευρά σας. Ήδη δεσμεύτηκα να απαντήσω στα ερωτήματά σας και θέλω να δραθώ της ευκαιρίας να το πράξω. Θα ήθελα να δώσω μια σύντομη επισκόπηση για το τι συμβαίνει σε σχέση με την διαδικασία Kimberley και ομάδες και ε, ομάδες ε, από βιομηχανικούς κύκλους συμμετέχουν στην ε, εποπτεία για την αποτελεσματικότητα του συστήματος πιστοποίησης και τεχνική συνδρομή και διοικητική συνδρομή θα παρέχεται από πλευράς τους στη διαδικασία Κέμπερλι. Αληθεύει ότι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών ήταν επικεφαλής το 2011. Ωστόσο θα ήθελα να προσθέσω εδώ κάτι ότι ήταν ένας από τους 12 εκπροσώπους ε, στη διαδικασία αυτή, Κίμπερλι, από πλευρά της κοινωνίας των πολιτών. Και οι άλλες 11 ΜΚΟ αμέσως επαλήθευσαν ότι δεσμεύονται σε σχέση με αυτή τη διαδικασία από πλευρά της κοινωνίας των πολιτών. Οι ΜΚΟ αυτές συμπεριλαμβάνουν μια Γερμανική Ένωση, μια Καναδική Ένωση Σύλλογο και οι υπόλοιποι είναι από την Αφρική. Αν μου επιτρέπετε σύντομα να αναφερθώ στο σχόλιο του σκιώδου του, επιτρέψτε μου μια παρατήρηση στη διαδικασία Κέμπελη. Γενικά ότι είναι κάτι πολύ λειτουργικό και αποτελεσματικό στον εθελοντικό χαρακτήρα που έχει, ώστε να μπορέσουμε από το 15% να πορευθούμε και να φτάσουμε στο 1%. Υπάρχουν όμως και κάποια όρια τα οποία δεν θα είναι δυνατόν να ξεπεράσουμε. Πάντα θα είναι εθελοντικού χαρακτήρα και σε σχέση με την συμμετοχή και την εφαρμογή όλων αυτών από πλευράς των εθνικών αρχών. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και πάλι ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα τώρα από πλευρά μας εξέταση σχεδίου έκθεσης, της δικής μου δηλαδή έκθεση το Νοέμβριο. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών, δύο ημέρες ε, ύστερότερα, ψήφιση προσέγγισης στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή το Δεκέμβριο και μετά στην Ολομέλεια θα περάσουμε προσέγγιση ίσως κατά την περίοδο συνόδου του Ιανουαρίου. Έτσι δεν νομίζω ότι θα είναι ε, μια οποιαδήποτε, δεν δημιουργείται κάποια καθυστέρηση για την εξέταση του χαρτοφυλακίου. Περνάμε στο σημείο 9. Πώς έχουν τα πράγματα σε σχέση με τις εξελίξεις του γύρου της Ντόχα του ΠΟΕ. Κατάσταση πρόοδου σχετικά με το αναπτυξιακό πρόγραμμα Ντόχα. Α, συγγνώμη, εδώ αγνόησα το 8. Το ξεπέρασα πηγαίνοντας υπερβολικά γοργά. Το 8 λοιπόν πρώτα. Επανερχόμαστε στο 8. Εξυγχρονισμός της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΕ Μεξικού. Εξέταση του αιτήματος προφορικής ερώτησης με απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως γνωρίζετε οι μεξικανικές αρχές, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, τον επικεφαλής του εκτελεστικού από πλευράς του προεδρικού συστήματος που ισχύει στο Μεξικό, υπήρξε ενδιαφέρον να εξυγχρονιστούν τα κεφάλαια της ε, ε, εταιρική σχέσης και συμφωνίας και ε, συνεργασίας Μεξικού ΕΕ από τη δεκαετία του 90 αυτή η συμφωνία που τον, τον Οκτώβριο 2000 άρχισε να ισχύει αυτό το θέμα λοιπόν εξετάστηκε, έγινε ένα ιδιαίτερα επίκαιρο και φλέγον θέμα για τους Μεξικανούς και αυτό επειδή είναι μία από τις ε, πρώτες συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και χωρών της Λατινικής Αμερικής από την Χιλή και σε σχέση με τις ε, σύγχρονες ε, συμφωνίες βλέπουμε ε, ότι υπάρχουν ε, κάποιες ε, διαφορές και μια και είναι τμήμα της ναύτα το Μεξικό, της Βορειοαμερικανικής Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου και με τον Καναδά και υπάρχει εδώ η συμφωνία αυτή που έχει ευρύτατα πλαίσια για τις επενδύσεις και το εμπόριο με τη ΣΥΠΑ και τον Καναδά θα πρέπει να υπάρξει μια συμμετρική ας το πω έτσι παράμετρο σε σχέση με τη συμφωνία που ισχύει μεταξύ Μεξικού ΕΕ ώστε να μην έχουμε, ας το πω έτσι, ένα μη επικαιροποιημένο και μη αποτελεσματικό πλαίσιο και να ανταποκρινόμαστε στις ε, υψηλές φιλοδοξίες που πρέπει να μας εμπνέουν. Οι Μεξικανοί από, την πλευρά, από πλευρά τους έχουν ε, εκφράσει και το ενδιαφέρον τους να εμπλακούν και να συνδεθούν με τη Συμφωνία Επενδύσεων και Εμπορίου με τη ΣΥΠΑ, την Διατλαντική Συμφωνία ΕΕΙΠΑ, ώστε να μην αφαιθούν εκτός μιας ενός τέτοιου πλαισίου συμφωνίας και να μην, ας το αγνοηθούν τα συμφέροντά τους. Κατά την τελευταία συνάντηση της μικτής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας ΕΕ Μεξικού στην πόλη του Μεξικού τον Ιούνιο εξέφρασαν και οι δύο πλευρές την επιθυμία τους να εμβαθύνουν περισσότερο σε αυτά τα θέματα αυτών των κεφαλαίων αμοιβαία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαφώς ανέφερε ότι υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί σε σχέση με την ε, διεύρυνση αυτών των ε, θεμάτων και η φιλοδοξία για μια αναθεώρηση πρέπει να είναι ευρύτερη και να επιτρέπει αμφωτέρωθεν τη δυνατότητα να εμβαθύνουμε στις σχέσεις εμπορίου μεταξύ μας σε σχέση με τις συμφωνίες με το Μεξικό από πλευράς ΕΕ που θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τη νέα γενναία συμφωνιών που ισχύει σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν για όλους αυτούς τους λόγους τι αποφασίσαμε. Αποφασίσαμε να υποβάλουμε μια προφορική ερώτηση με, που θα απαντηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Κούτας είναι ο ε, εισηγητής μας για αυτά τα θέματα. Και έχει τον λόγο κύριε Κούτα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, περιγράψτε πολύ σωστά την κατάσταση. Στη σχέση μας τώρα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Μεξικό η παρουσία στιγμή είναι σημαντική. Δεν πρέπει να χάσουμε την ορμή αυτών των διαπραγματεύσεων. Διότι προφανώς ό,τι αποφασίσουμε και ό,τι επιτευχθεί εν τέλει στο TTIP θα επηρεάσει επίσης και τη συμφωνία με το Μεξικό. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να αναλάβει μια στάση και να επιμείνει σε μια πιο φιλοδόξη συμφωνία τονίζοντας κάποια σημεία και ζητώντας κάποιες διευκρινήσεις από την Κομισιόν. Κατά την απόψή μου, πολύ σημαντικό είναι να συμπεριληφθεί ένα κεφάλαιο βιώσιμης ανάπτυξης με μια ρήτρα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το σχετικό μηχανισμό, όλα αυτά έχουν υλοποιηθεί ήδη στη Συμφωνία με την Κολομβία. Πιστεύω επίσης ότι είναι σημαντικό η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κολομβίας να αποτελέσει ορόσημο για μελλοντικές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω επίσης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εκφράσει την απόψή της όσον αφορά τις συνέπειες του εξυγχρονισμού της συμφωνίας για την πολιτική συνοχή, των περιβάλλον καθώς και τους τρόπους βελτίωσης των κεφαλαίων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, θα ήθελα να ενημερώσω όλες τις πολιτικές ε, ομάδες. Ε, θα ήθελα μάλλον να τις ευχαριστήσω για τη συμβολή τους και για να συμφωνήσουμε όλοι, γιατί υπάρχουν κάποιες διχογνωμίε αυτή τη στιγμή, θα διοργανώσω μια συνάντηση, όπου ελπίζω να επιτευχθεί συμβιβασμό μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων. Στο μεταξύ, προτείνω να δώσουμε προσοχή στο να κατανοήσουμε πού υπάρχουν τα προβλήματα, για ποιες ομάδες και ενδεχομένω να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κάποιες συμβιβαστικές ε, στην συνάντηση που θα λάβει χώρα. Ευχαριστώ. Ε, από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα. Θέλω να υποστηρίξω αυτό το οποίο αναφέρθηκε από τον συνάδελφο. Υπάρχει και από τις δύο πλευρές η ανάγκη να εμβαθύνουμε σε σχέση με, το, με τις εμπορικές σχέσεις. Πράγμα το οποίο θα έδινε την δυνατότητα να ευθυγραμμιστούμε με μια νέα συμφωνία νέας γενεάς εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Μεξικού αληθεύει ότι παρότι υπάρχει αυτή η κοινή βούληση, δεν υπάρχουν συγκλήσεις ε, για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτή, αυτός ο εξυγχρονισμός. Ένα σχέδιο λοιπόν ερώτησης ε, προς το, το, από πλευράς του κύριου Κούτας. Θέλω να τον συγχαρώ για αυτό το εγχείρημα είναι θετικό για να επικεντρωθούμε στα εμπορικά θέματα και να δούμε ποιε είναι οι απόψει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εμβάθυνση των εμπορικών μα σχέσεων το δυνατόν νωρίτερα με το Μεξικό. Ευχαριστούμε. Έχετε και την προφορική ερώτηση στο αρχείο σας. Ακολουθεί με την Κάζα ναι, Κρυπτοάλντε. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω ότι είμαστε γενικά ικανοποιημένοι με την προφορική ερώτηση που προετοίμασε ο συνάδελφος κ. Κουτάς. Πιστεύω ότι τα σημαντικότερα ζητήματα περιλαμβάνονται. Πράγματι σε αυτή την ερώτηση τονίζοντας ιδιαίτερα την ανάγκη δεσμευτικού κεφαλαίου αηφόρου ανάπτυξη με τη συμπερίληψη μιας ρήτρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιστεύω ότι αυτό είναι σημαντικό για μια χώρα όπω το Μεξικό. Επίσης ε, φυσικά είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που βλέπουμε ότι αναφέρεται ότι θέλουμε να δούμε πώς προτίθεται να δράσει η Κομισιόν όσον αφορά το κεφάλαιο για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ώστε να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα η νομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η φοροδιαφυγή πολύ σημαντικά ζητήματα πιστεύω στο πλαίσιο λοιπόν των διαπραγματεύσεών μας ε, θα αξιοποιήσουμε και τη συμφωνία TTIP με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Καλό θα ήταν λοιπόν να, στη συμφωνία αυτή, στις διαπραγματεύσεις για το TTIP, να συμπεριλάβουμε και αυτή, να αναφέρουμε και αυτήν εδώ τη συμφωνία. Αναμένουμε την απάντηση στις ερωτήσεις από την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε η ΣΥΑΡ. Κυρία Κλάρκιν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα για τις εμπορικές σχέσεις με το Μεξικό. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα επίκαιρο το ζήτημα αυτό, καθώς εξελίσσονται και οι διαπραγματεύσεις TTIP. Καλό είναι λοιπόν που ενημερώνουμε τις σχέσεις με εταίρους όπως το Μεξικό. Είχα μια συζήτηση με την πρέσβερα του, την απερχόμενη πρέσβερα του Μεξικό και μας είπε ότι πρέπει να συμπεριλαμβούμε όλους τους εταίρους ε, και να συμφωνήσουμε μαζί τους και να παρέχουμε συνοχή στις διαπραγματεύσεις μας ε, όσον αφορά τις διευθετήσεις ειδικότερα με έναν εταίρο όπως το Μεξικό που είναι επίσης και γείτονα ε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή είναι η απόψή μου και ανυπομονώ για τις επόμενες συζητήσεις. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστούμε, Σκάκελε. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το προσχέδιο αυτό με το οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε σε άλλες γραμμές και εμείς ε, προσβλέπουμε σε μία συνάντηση για αυτό το θέμα γιατί υπάρχει κάτι ακόμα το οποίο θα θέλαμε να προσθέσετε και ανέφερε και ο άλλο Φεζάκ αφορά ε, το κεφάλαιο για τις ε, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Ε, ξέρουμε το προηγούμενο προσχέδιο ότι η Επιτροπή θα εξέταζε το θέμα για το πώς ένα τέτοιο κεφάλαιο θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση. Όμως, πρέπει να διευκρινίσουμε προς ποια κατεύθυνση θέλουμε να κινείται αυτή η βελτίωση. Προς τα πού θα πρέπει να κινηθεί η Επιτροπή, κατά τη γνώμη μας και συμφωνώ ότι το κεφάλαιο περί χρηματοοικονομικών ε, υπηρεσιών ε, θα πρέπει να επιλύσει ζητήματα ξεπλήματος χρήματος γιατί διακόπτει ο Πρόεδρος, ε, να αναφερθούμε στις, στην ακριβή διατύπωση για να σταματήσει το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εκτός μικροφώνου το σχόλιο. Okay. Συνεχίστε. Ναι, αυτή είναι η πρώτη αλλαγή που θα θέλαμε να ζητήσουμε. Αλλά συμφωνούν όλοι, φαντάζομαι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να επαναλάβω τόσο, όσα συνάδελφοι. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εκπόνηση της ερώτησης και συμφωνώ με τη γενική προσέγγιση. Να προσθέσω μόνο ένα σημείο, το οποίο είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου, ε, για το κεφάλαιο περί ε, Νομίζω ότι πραγματικά θα πρέπει να προσθέσουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών. Ίσως αυτό μπορεί να συζητηθεί κατά αυτή τη συνάντηση, γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και αν δείτε τη σύγκληση μεταξύ και την οριζόντια διασύνδεση μεταξύ των ε, συμφωνιών του ΣΥΤΑ και το καθεξής, όλα αυτά φαίνονται όμως. Υπάρχουν και διαπραγματεύσεις σε TTP που σίγουρα θα επηρεάσουν και τις εμπορικές μας σχέσεις με το Μεξικό. Πρέπει να είμαστε λοιπόν όσο πιο συγκεκριμένοι γίνεται. Συνάδελφε, μπορούμε να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει με ε, την ε, επίλυση διαφορών και αυτό εντάσσεται και στο κεφάλαιο επενδύσεων. Οι συμφωνίες επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ θα αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες διμερείς ε, συμφωνίες με τους εταίρους και στην προκειμένη το Μεξικό πώς μπορούν οι δικές μας επιχειρήσεις να συμφωνήσουν, να αντεκατασταθούν οι συμφωνίες επενδύσεων όταν υπάρχουν τέτοιοι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών από Ευρωπαϊκή Συμφωνία που δεν προβλέπει τέτοιο μηχανισμό. Μπορείτε να μου το απαντήσετε. Από μόνο σας, ε, μέσω του ερωτήματός σας, γιατί αν καταλήξουμε σε μια τέτοια συμφωνία, ε, με μηχανισμό επίλυση διαφορών από, μεταξύ δύο κρατών, απαντάτε το ερώτημά σας. Επομένω, αυτό πρέπει να συζητήσουμε μαζί και με την Ευρωπαϊκή και το Συμβούλιο είναι πώς μπορούμε να οργανώσουμε αυτές ε, τις ε, συμφωνίες επενδύσεων με τρίτες χώρες που περιλαμβάνουν και τον κανονισμό του ΠΟΕ. Πρόεδρος, αυτό σημαίνει ότι χωρίς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών δεν υπάρχουν ε, συμφωνίες ε, επενδύσεων. Θα μείνουμε δηλαδή με τις διμερείς ε, και μόνο συμφωνίες επενδύσεων, γιατί μόνο εκεί υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί. Από την Επιτροπή, κανείς. Ποιος εκπροσωπεί την Επιτροπή για αυτό το θέμα. Ζόρις Τουρίνο, από την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Βιτορίνο, από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Δυστυχώ, ο συνάδελφός μα από τη Γενική Διεύθυνση αρρώστησε, ασθένησε και δεν μπόρεσε να παραστεί και για την που παρακολουθεί και τις εμπορικές σχέσεις με το Μεξικό. Είναι ελεύθερη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να πει ποιος θα παρέμβει από τα μέλη. Λοιπόν, σημειώσαμε φυσικά τα σχόλια τα οποία έγιναν από πλευράς ε, των συμμετεχόντων για το κεφάλαιο και για την αηφορό ανάπτυξη που ήταν και η ας το πω έτσι ένδειξη ότι δεν είχε αυτό ε, τον πιο αποτελεσματικό, το πιο αποτελεσματικό πλαίσιο σε σχέση με το Μεξικό και τα όσα αναφέρθηκαν σε σχέση με την ε, επικαιροποίηση, σε σχέση με συμφωνίες που έχουμε υπογράψει. Και για το θέμα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών φυσικά σημειώσαμε τα σχόλια τα οποία έγιναν και την διασύνδεση με το πλήσιμο ξέπλυμα χρήματος και είναι κάτι το οποίο σε σχέση με τη συμφωνία με την Κολομβία και το Περού ισχύει και φυσικά θα πρέπει να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε σχέση με τις συμφωνίες ΕΕ επί συναφών θεμάτων και εμπορίου. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτά από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τώρα ας επανέλθουμε στον εισηγητή μας κύριο Κούτας θετική η ανταπόκριση. Έτσι, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους. Όπως είπα, θα προσπαθήσω να διοργανώσω μία συνεδρίαση ώστε να έχουμε τις διαφορές που υπάρχουν και όλοι να μπορέσουν επ' αυτών να τοποθετηθούν για να διευθετηθούν. Και σε σχέση με τα όσα αναφέρθηκαν θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η καλύτερη διατύπωση που θα υιοθετηθεί ώστε όλες οι ομάδες να ικανοποιηθούν και δεν βλέπω για ποιον λόγο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποια προσχήματα. Πρέπει όλοι να μπορέσουν να ενταχθούν. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την προφορική ερώτηση αναμένω όπως και ανέφεραν και όλοι οι συνάδελφοι ότι θα έχουμε μια πολύ θετική τοποθέτηση και απάντηση για αυτήν την ερώτηση. Είναι πολύ σημαντικό για τα θέματα εμπορίου ΕΕ και Μεξικού αυτό. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ καλή η συζήτηση. Χρονοδιάγραμμα. Η μετάφραση για τις έκθεσεις 25η του μήνα ψήφιση στην Επιτροπή μας 14η Οκτωβρίου. Τώρα το θέμα, το ζήτημα 9 η πρόοδος που έχει συμμεθεί με το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ντόχα και για πρόταση ε, ψηφίσματος το σχέδιο ψηφίσματος είναι διαθέσιμο στα χαρτοφυλάκια σας, στους φακέλους σας. Είμαι εισηγητής εγώ προσωπικά και θα συμμετέχουν και προσυπογράφουν και συνάδελφοι ως και συμπρόεδρος της ε, ομάδας ε, από πλευράς ε, του Ευρωκοινοβουλίου για τον ΠΟΕ. Στο σχέδιό μας λοιπόν έχουμε τονίσει και πάλι τη δέσμευσή μας στην πολυμερή προσέγγιση, στην πολυμερή ημερήσια διάταξη από πλευράς ΠΟΕ και είναι, θα έλεγα, κέρια σημασία, πολύ σημαντικό να αποσταλεί ένα ισχυρό και σαφές μήνυμα από το Ευρωκοινοβούλιο σε σχέση με αυτό το θέμα, αποσαφηνίζοντας τα πράγματα και λαμβάνοντας υπόψη το ότι χρειαζόμαστε και πρέπει να έχουμε να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο σε σχέση με τον Μπαλί κατά τα τέλη, μέχρι τα τέλη του έτους και για τα θέματα της ανάπτυξης, της Επιτροπής ε, Ανάπτυξης ε, έχουν και αυτά ληφθεί υπόψη ώστε να ε, εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Για το, τη δέσμη μέτρων για το Μπαλί που ευελπιστούμε ότι θα μπορέσει να ολοκληρωθεί οι συζητήσεις για τα μέσα και τη διευκόλυνση για το εμπόριο δεν ακολουθούν την ταχεία πρόοδο που προβλέπαμε και είχαμε επιθυμήσει, δεν θα ονοματίσω και δεν θα κατηγορήσω κανένα. Αναφέρουμε σε σχέση με το ψήφισμα ότι θα πρέπει αυτό το μέσο να αποβεί προς όφελος ε, και των ε, αναπτυσσομένων χωρών, θίγει θέματα σε σχέση με την συμφωνία και τα θέματα προμηθειών και για την συμφωνία για την, τις τεχνολογίες και πολυμερή χαρακτήρα που πρέπει να έχουν οι δεσμεύσεις μας μέσα στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών. Ας έχουμε λοιπόν την δυνατότητα να παρέμβουν οι σκιώδεις εισηγητές. Ο συνάδελφος που είπαμε δεν παρίσταται. Κάποιος που θέλει να λάβει τον λόγο, παρακαλώ. Παύλο Γαρθάτη, Από την Επιτροπή, παρακαλώ εσύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να δώσουμε και τη δική μας άποψη επί του ζητήματος. Αρχικά να ευχαριστήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το σχέδιο ψηφίσματος. Θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα ε, πολύ καλό κείμενο και είμαστε βεβαίως και διατεθειμένοι να συνεργαστούμε μαζί σας όπως πάντα. Να συμβάλλουμε και εμείς σε αυτό το ψήφισμα. Για την έκθεση που έχετε αυτή τη στιγμή στη Γενέβη βρισκόμαστε ε, σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις. Έχουμε τον νέο Γενικό Γραμματέα που ξεκίνησε από τις ε, αρχές Σεπτεμβρίου. Ήδη έχει διοργανώσει πολλές ε, ε, συναντήσεις σε επίπεδο πρέσβεων για να δούμε αν και κατά πόσο μπορούμε να έχουμε τα θετικά αποτελέσματα που όλοι επιθυμούμε στο Μπαλί στα τέλη του έτους. Να τονίσω μόνο δύο ζητήματα. Όχι μόνο θα έχουμε την Συμφωνία Διευκόλυνσης Εμπορίου ως βασικό ε, σημείο και στοιχείο του πακέτου του Μπαλί. Αυτό λοιπόν δεν θα ήταν μόνο εποφελές για τους δικούς μας εισαγωγής και εξαγωγής, αλλά και για τις αναπτυσσόμενες χώρες και το εμπόριό τους. Επίσης το να έχουμε ένα τέτοιο θετικό αποτέλεσμα στο Παλί θα δείξει ότι ε, η ε, πολυμερής ατζέντα διαπραγματεύσεων εξακολουθεί να υφίσταται και αυτό είναι κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τους διαπραγματευτές στη Γενέβη. Πέρα λοιπόν των τεχνικών αποτελεσμάτων που θα έχουμε επιτάπητος και μια συστημική προσέγγιση σίγουρα θα ε, αποτελέσει κινητήρο μοχλό των προσπαθειών μας στη Γενέβη. Πράγματι, οι διαπραγματεύσεις για τις ε, εμπορικές διευκολύνσεις δεν έχουν προχωρήσει όσο θα έπρεπε. αλλά μπορούμε να τα καταφέρουμε. Όπως πάντα βέβαια αυτά τα πράγματα είναι αλληλένδετα. Εδώ έχουμε τις διαπραγματεύσεις ε, στα γεωργικά ζητήματα που σχετίζονται και με την ασφάλεια τροφίμων στην Ινδία. Είναι κέριο σημείο αυτό. Είδατε και τις ε, τελευταίες ε, εβδομάδες τις διαταραχές και στο πολιτικό επίπεδο στην Ινδία για που καλούν, ε, απευθύνουν έκκληση για την ε, σωστή εφαρμογή ε, του, της νομοθεσίας για την ασφάλεια τροφίμων, όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν καλές προοπτικές σε σχέση με το παρελθόν. Ίσως αυτό το ανέφερε και αξιωματούχος επειδή ακριβώς έφευγε και αγκατέλειπε τη θέση του, όμως έχουμε την αίσθηση ότι είναι κάτι το εφικτό και σίγουρα η Επιτροπή, υπό και τη δική σας ε, ε, καθοδήγηση, στην Επιτροπή λοιπόν κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να έχουμε μια δέσμη που θα είναι θετική για τους εξαγωγείς μας, για την ανάπτυξη και θετική και για τον ε, Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Γιατί τη σήμερα ημέρα αυξάνεται ο προστατευτισμός και έτσι χρειαζόμαστε έναν ισχυρό ΠΟΕ για να προσέχει εντό εισαγωγικών και το παγκόσμιο εμπόριο και την παγκόσμια οικονομία. Σα ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σα για ερωτήσει. Είστε αισιόδοξο. Πείτε μα με ειλικρίνεια, δεν θα το πούμε σε κανέναν. Πάντα είμαι αισιόδοξο στη ζωή. Συγγνώμη που είναι προσωπική η δήλωσή μου. Είμαι αισιόδοξο. Έχουμε ένα νέο γενικό διευθυντή Βραζιλιάνο. Θα πάμε στην Ινδονησία, στο Μπαλί. Δεν θα πάμε στο Μπαλί για να αποτύχουμε. Ήδη αποτύχαμε στη Γενέβη. Το πιστεύω ότι θα πετύχει και πιστεύω ότι ως διαπραγματευτές είναι σημαντικό να έχουμε αυτοπεποίθηση για αυτό που κάνουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Δεν είμαι αγαθός, γνωρίζουμε τους κινδύνους που υπάρχουν όπως έχουμε πει σχετίζονται με την εγχώρια ατζέντα ορισμένων εταίρων αλλά σίγουρα η Κομισιόν κάνει ό,τι μπορεί για να διευκολύνει την επίτευξη αποτελέσματος και για τους τρεις πυλώνες, διευκόλυνση των συναλλαγών, γεωργία και τα αναπτυξιακά ζητήματα ειδικότερα όσον αφορά τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα γίνουν προσπάθειες οι οποίες θα καταλήξουν σε επιτυχές αποτέλεσμα. Το πρόβλημα είναι κατά πόσο έχουμε απαραίτητους πόρους για να πείσουμε σε χώρες αντιστέκονται ακόμα. Αυτές που ακόμα δεν έχουν πιστεί ή που σε κάθε περίπτωση αναμένουν κάποιο ικανή ανταμοιβή για το κοινοβούλιο. Για μας είναι σημαντικό, διότι πίστευω ότι δεν πρέπει να μην διαφανεί καμία αμφιβολία ότι υπερασπιζόμαστε το διμερές σύστημα συναλλαγών στον ΠΟΕ και δεύτερον γιατί θα διοργανώσουμε μια συνεδρίαση, μια διακοινοβουλευτική συνεδρίαση μαζί με την Υπουργική Διάσκεψη στον Παλή είναι σημαντικό αυτό για μας στο Κοινοβούλιο. Αυτό διότι εμείς ε, συμβάλλουμε όχι μόνο στην προβολή του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος και των εμπορικών κανονισμών και τη ε, ρύθμιση του εμπορίου, αλλά θέλουμε να δείξουμε ότι και εμείς ως Κοινοβούλιο εμπλεκόμαστε σε εμπορικά ζητήματα. Θέλουμε κάθε Κοινοβούλιο να είναι όσο δραστηριόμαστε εμείς στην εμπορική πολιτική ενώπιον των κυβερνήσεων μας. Ε, ε, ευχαριστώ που προτείνετε αυτό το ψήφισμα. Παρότι αν δεν κάνω λάθος είχε υπάρξει ένα άλλο ψήφισμα στην Τόχο που είχαμε πει ότι τώρα χρειαζόμαστε μια νέα λύση καινοτόμο και έτσι έχω βουλήσει κατά πόσο θα βρεθεί κάτι τέτοιο στον παλί. Ας πάμε και βλέπουμε. Πιστεύω ότι το θετικό κομμάτι σε, αυτή την, σε αυτό το ψήφισμα είναι ότι έχουμε νέα γλώσσα, χρησιμοποιούμε νέα γλώσσα ώστε να προσφέρουμε κάτι ενδιαφέρον και για τις αναπτυσσόμενες χώρες και εκεί θα πρέπει να εστιαστούν οι διαπραγματεύσεις. Από αυτή την άποψη δεν μας ικανοποιούν ιδιαίτερα οι παράγραφοι 9 και 11 διότι εμείς οι πράσινοι δεν καταλαβαίνουμε πώς τέτοιες πρωτοβουλίες ε, μπορεί να συμβάλλουν επικοδομητικά για τις, ε, και υποφελώς για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης απορρίπτονται από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Δεν είμαι λοιπόν βέβαιη κατά πόσο κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ενταχθεί στο όλο πλαίσιο. Επίσης στην παραγράφο 7 για τη Γεωργία αυτό ήταν ένα κομβικό σημείο και πιστεύω ότι εδώ δεν αναφέρονται νέα βήματα τα οποία θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν για να επιτευχθεί κάποιο αποτέλεσμα. Επίσης, για την απόψή μου, δεν είναι σαφές ε, αν θα μπορούσε σύντομα να υλοποιηθεί κάποιο πακέτο διευκόλυνσης του εμπορίου. Αν κάνω λάθος, παρακαλώ, ενημερώστε με εφόσον υπάρξει πακέτο διευκόλυνσης των συναλλαγών δεν βλέπω ποια ακριβώς θα ήταν η παρακολούθηση ώστε να επιτευχθεί πλήρης ανάπτυξη των όσων συμφωνήθηκαν στο γύρο της Δόχα. Ίσως θα μπορούσε η Κομισιό να μας διαφωτίσει επί αυτού. Εγώ διατηρώ ενδιασμούς. Έχω επιφυλάξει κατά πόσο θα δούμε κάτι νέο στον Παλί. Ωστόσο είναι σημαντικό να εστιαστούμε στην επίτευξη νέων βημάτων σημαντικών για την ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών και την ικανοποίηση των αναγκών των χωρών αυτών και των πληθυσμών τους. Θα αναμένουμε τις τροπολογίες σας. Άλλο έτοιμο, Νικολό Ρινάλντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες θα ήθελα να πω για να βελτιώσουμε το σχέδιο ψηφίσματος παρότι είναι σίγουρα ευρύτερο και αποδεκτό αυτό το ψήφισμα. Θα θέλαμε όμως να συμπεριληφθούν και κάποια θέματα όσον αφορά τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προαγωγή της πολυμερούς προσέγγισης στο γύρο της Ντόχα για καλύτερες προοπτικές ε, όσον αφορά την ενίσχυση για παράδειγμα της κοινοβουλευτικής διάστασης ε, δεν είναι το πρόβλημα της ε, έλλειψης, της απουσίας ηγετικού ρόλου από πλευρά Κοινοβουλίου. Το θέμα είναι το να υπάρχουν κάποιοι να ακολουθήσουν. Ναι, είναι κέρια σημασία αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε και για τους υπόλοιπου. Επίσης, και στην τροπολογία μα θα υπάρχει κάποια αναφορά, διότι δεν γίνεται αυτό εδώ, για την ανάγκη να υπάρχει φορολογική η δικαιοσύνη και ισότητα, καταπολέμηση τη διαφθορά δυνατότητα ενίσχυση ε, τη απλούστευσης είναι αυτά θέματα τα οποία πρέπει να βαίνουν εκ παραλίλου με την διευκόλυνση και τις δυνατότητες που θα διαμορφώσουμε για το εμπόριο και τι εμπορικές συναλλαγές. Επίσης θα προσπαθήσουμε να τροποποιήσουμε την παράγραφο 9 μετά από τα όσα μόλις είπε η Φρανσίσκα ώστε να καταφέρουμε να καταστήσουμε σαφέ ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίσουν τους εθνικούς στόχους στις πολιτικές τους όσον αφορά την απελευθέρωση των δημόσιων υπηρεσιών και να μην υπάρχει, ας το πω έτσι, κάποιος περιορισμός ή ε, ε, περιστολή όσον αφορά αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Εσείς ε, κύριε Νίκολα από την ΓΚΟΕ σας ευχαριστώ. Συμμερίζομαι τις απόψεις των συναδέλφων και θέλω να ευχαριστήσω για τη σύνταξη αυτού του κειμένου. Έχουμε αρχίσει να συζητούμε αυτά τα θέματα και σε σχέση με τα θέματα περιφερειακής ανάπτυξης και όσον αφορά και τα θέματα του ΠΟΕ και την ε, δυνατότητα να εμπλακούμε σε αυτά. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα του ψηφίσματος. Νομίζω δίνεται μια πραγματική εικόνα δίνοντας τις προκλήσεις που παρουσιάζονται σε σχέση με ένα πολυμερές πλαίσιο. Αλλά θα ήθελα να προχωρήσουμε και πιο πέρα. Αν δεν υπάρξει συμφωνία σε σχέση με το γύρο της Ντόχα, το θέμα της απεσιοδοξίας ε, το οποίο αναφέρθηκε πώς θα αντιμετωπιστεί αν δεν θέσουμε σαφώς ε, τις ε, ευθύνες από πλευράς μας ε, όσον αφορά την Τόχα, το γύρο της Τόχα. Ποιες είναι οι ε, ευθύνες, ε, ποια ευθύνη έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το ένα ή άλλο θέμα. Και φυσικά αυτό αφορά εμάς ιδιαίτερα και θα ήθελα να πω ότι στο άρθρο 3 παράδειγμα με πολύ καλό τρόπο περιγράφεται το πού βρισκόμαστε και ποιες είναι οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δεν θα πρέπει όμως να πούμε ότι είναι ένα αναγκαίο μέσο, αλλά είναι ένα μέσο να συνδέσουμε την πραγματικότητα σε σχέση με τα κράτη-μέλη και τον ΠΟΕ με την δυνατότητα να συμμετέχουν και να παρακολουθούν τα θέματα αυτά στον ΠΟΕ. Αν προσθέσουμε τέτοια θέματα σε σχέση με το ψήφισμα μπορούμε στην κοινοβουλευτική δομή και στην δυνατότητα να προχωρήσουμε κοινοβουλευτικά θα είχαμε μια πολύ σημαντική συνεισφορά. Ευχαριστώ. Εσείς παρακαλώ. Εσείς παρακαλώ από την Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Απλά σύντομα να αναφερθώ σε κάποια από τα θέματα και τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Πώς ε, το μέσο διευκόλυνσης του εμπορίου θα διευκόλυνε τα ε, υπόλοιπα όσον αφορά την προαγωγή τους. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αυτή η συμφωνία μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο θα άνοιγε την πύλη για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Τώρα, για το αν μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή η δυνατότητα θα ήταν καλό. Αν όχι, θα ήταν δύσκολο να δει κανεί ποιε δυνατότητες θα υπήρχαν στο μέλλον. Τώρα, θα πρέπει να είναι, αναφέρθηκε, καλό, θετικό για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ένας από τους λόγους για τους οποίους είναι δύσκολο να ολοκληρωθεί αυτό το εγχείρημα είναι να διαφοροποιηθούμε μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών και ε, ε, των αναπτυσσόμενων χωρών και των ανεπτυγμένων χωρών. Δεν είναι τα ίδια σε σχέση με 20 χρόνια πριν οι, ε, οι, οι ανάγκες ε, για τις αναπτυσσόμενες χώρες ε, ε, αναπτύσσονται σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Θα ήταν σημαντικό λοιπόν και σας παρακαλώ να εμβαθύνετε σε αυτό, να υπάρξει μια επιλογή μιας ε, ε, μεταβατικής περίοδου προτού υπάρξει δέσμευση μέσα σε αυτό το πλαίσιο αυτής της συμφωνίας. Αυτό θα ήταν ένα βήμα προς την κατεύθυνση να υπερβούμε, να ξεπεράσουμε τα εμπόδια. Αναφέρθηκε το θέμα της διαφθοράς. Οι ε, διατάξεις ε, σε σχέση με τις κυρώσεις ε, και τα πρόστιμα τα οποία θα μπορούσαν να επιβάλλονται όσον αφορά περιπτώσεις διαφθοράς είναι σίγουρα μια από τις δυσκολίες που αναφύονται. Ο, ρόλος του Κοινοβουλίου και η παρατήρηση φυσικά είναι κάτι το οποίο πάντα υποστήριζε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα προσπαθούμε και στον Παλί επίσης να ε, καθορίσουμε και τη δυνατότητα συμμετοχής των εκπροσώπων ε, του Κοινοβουλίου στις, ε, στις, διαπραγματεύσεις του, στον Παλί ώστε να μπορούν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και εν τέλει, εν κατακλείδη, δεν είναι πανάκια το εμπόριο φυσικά. Επίσης πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποια ας το πω έτσι τάση που να ε, διανοίγει μια άλλη προοπτική για το εμπόριο. Δεν θέλω να αναφέρω ότι κάποιοι είναι υπεύθυνοι μετά από τα τόσα χρόνια διαπραγματεύσεων. Είναι κάτι το οποίο είναι φυσικό και συνεχίζουμε να καταβάλουμε προσπάθειες λαμβάνοντας υπόψη την ε, πολιτική υποστήριξη που πρέπει να απορρέει για ένα πολυμερές ε, ε, τέτοιο εμπορικό πλαίσιο και σε τακτά διαστήματα τα μέλη του ΠΟΕ θα μπορούν να, μπορούν να παρεμβαίνουν ώστε να προχωρήσει αυτό το χαρτοφυλάκιο. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ. Και αυτό ολοκληρώνει αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων, την πρώτη συζήτηση. Κατάθεση τροπολογιών ως προθεσμία η 19η Σεπτεμβρίου στις 18.00 το απόγευμα ψήφιση προσέγγιση στην Επιτροπή μας τον Οκτώβριο. Προσβλέπω στην κατάθεση τροπολογιών από πλευρά σας. Το θέμα υπαριθμών 10 τώρα στην ημερήσια διάταξη που ακολουθεί είναι ο αντίκτυπος των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες, τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με τρίτες χώρες όσον αφορά το πλαίσιο της Τελωνιακής Ένωσης και ιδίως εταίρους της ΕΕ, κυρίως στην Τουρκία. Όπως θα θυμόσαστε, τον Ιούνιο εφέτος είχαμε, ακούσαμε και την παρουσίαση που δόθηκε από ανώτερο εκπρόσωπο υπάλληλο του Υπουργείου Εμπορίου της Τουρκίας, ο οποίος μας εξέθεσε κάποια μελήματα, κάποιες ε, προσπάθειες όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ και τρίτες χώρες, ε, όπως για παράδειγμα της είπα. Σύμφωνα με την Τελωνιακή Συμφωνία, Τελωνιακής Ένωσης μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας, η Τουρκία θα υποστεί, ας το πω έτσι, τις επιπτώσεις επιπτώσεις της εμπορικής συμφωνίας, μιας εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών. Δηλαδή σε σχέση με προτιμησιακά καθεστώτα έναντι τρίτων χωρών, χωρίς χαρακτήρα αμοιβαιότητας. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα λοιπόν η Τουρκία να μπορέσει να αναπτύξει διαπραγματεύσεις με αυτές τις χώρες με τις οποίες διαπραγματευόμαστε εμείς, ώστε η Τουρκία να μπορεί να έχει και εκείνη πρόσβαση στις χώρες αυτές με ένα προτιμησιακό καθεστώς, διασφαλίζοντας έτσι την αμοιβαιότητα όσον αφορά τις εμπορικές της σχέσεις με τις χώρες αυτές. Αποφασίσαμε να τεθεί προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απάντηση η συγητής για αυτό το θέμα είναι ο Μέτιν Καζάκα. Με την έχει τον λόγο για να τοποθετηθεί επ' αυτού. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως αναφέρθηκε είχαμε μία ειδική δήλωση του τουρκικού Υπουργείου Οικονομίας για ε, τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει η Τουρκία λόγω των ε, διαπραγματεύσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ. Γι' αυτό και τον Ιούλιο οι διορμοτευτές αποφάσισαν να θέσουν ένα τέτοιο ερώτημα χωρίς ε, ψήφισμα για την εφαρμογή, τη συμμετοχή μάλλον της Τουρκίας και άλλων τέτοιων χωρών που δεν αποτελούν μέλους της Τελωνικής Ένωσης σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, τρίτες χώρες ε, για τέτοιες διαπραγματεύσεις για που αφορούν τα εμπορικά ζητήματα. Ξέρετε ότι η Συμφωνία Τελωνική Ένωση με την Τουρκία υποχρεώνει την Τουρκία να ακτιγραμμιστεί με ε, την Ευρωπαϊκή Κοινή ε, Εμπορική Πολιτική, με την εφαρμογή των ίδιων προτιμησιακών καθεστώτων ε, με τις τρίτες χώρες, αλλά η Τουρκία, εφόσον δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιτρέπεται να υποφεληθεί αυτών των προτιμησιακών εμπορικών καθεστώτων. Βεβαίως αυτή η ασύμετρη ε, θέση μπορεί να επηρεάσει και να έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην τουρκική οικονομία. Το 2010 υιοθετήσαμε δικό ψήφισμα για, την, ε, για τις ε, τελωνικές οικονομικές, εμπορικές και οικονομικέ σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση-Τουρκία, όπου είπαμε ότι αυτό το στοιχείο είναι πολύ σημαντικό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Τουρκία. Όμω, βλέπουμε ότι αυτή η ασύμετρη θέση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο στις σχέσεις μας, γιατί ιδίως για την Τουρκία, οι τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει ε, FTAs με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να έχουν ε, πρόσβαση στην αγορά χωρίς ποσοστώσεις, χωρίς δασμούς και χωρίς ε, αμοιβαιότητα. Ε, αυτό δεν ισχύει με ε, άλλους εταίρους όπως ε, η Ανδόρα και το Σαν Μαρίνο. Και δεύτερον, επειδή η Τουρκία έχει αντικειμενικές δυσκολίες κατά τη διαπραγμάτευση παράλληλων εμπορικών συμφωνιών με χώρες που έχουν ήδη de facto πρόσβαση στην αγορά του, της, λόγω της ύπαρξης της Ελληνικής Ένωσης. Για να επιλύσουμε λοιπόν αυτό το ζήτημα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας της Τουρκίας ε, ανέφερε διάφορες ε, πιθανές λύσεις ε, συμπεριλαμβάνοντα και κάποιε λύσει για την ενδεχόμενη εκπροσώπηση τη Τουρκία και άλλων εταίρων τη Τελωνική Ένωση κατά τη διαπραγμάτευση τέτοιων συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου με τρίτε χώρε και με την ύπαρξη της λεγόμενης ρήτρας, τουρκικής ρήτρας σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Όλα αυτά θα πρέπει να τα αναλύσουμε. Όμως προς το παρόν η προφορική ερώτηση ακόμα δεν έχει τύχει συμφωνίας ε, εφόσον συνεχίζονται οι συζητήσεις στις πολιτικές ομάδες για το πεδίο εφαρμογή ε, ε, του ζητήματος και πώς μπορούμε να λάβουμε υπόψη τις θέσεις όλων των εταίρων, γιατί διαφέρει η άποψη της Τουρκίας από των υπολείπων εταίρων της Τελωνιακή Ένωσης. Γι' αυτό και προτείνω να μην συζητηθεί ένα προσχέδιο, αλλά να συνεχίσουμε τις εργασίες μας επί ενός κοινού κειμένου και μετά να προτείνουμε ε, την υιοθέτηση της ε, συμπεφωνημένης προφορικής ερώτησης κατά την επόμενη συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει λοιπόν προσχέδιο προς το παρόν, όμως έχουν παρουσιαστεί κάποιες ιδέες από τους ε, εισηγητές. Σκιώδης. Ο Μπέρτ Λάγκε, πρόεδρε, πολύ σύντομα, υποστηρίζουμε την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή δεν έχουμε βέβαια λύση γι' αυτό. Κατά τούτο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητείται, καλείται να τοποθετηθεί και να εξετάσει διάφορες εναλλακτικέ δυνατότητες και να επιλέξει από αυτές. Πώς λοιπόν θα μπορούμε σε σχέση με την Τελωνιακή Ένωση να λάβουμε υπόψη εταίρους μας και κατά δεύτερον να δούμε τι θα μπορεί να γίνει με την ναύτα όσον αφορά τα θέματα του Μεξικού και μόλις πιο πριν είχαμε το θέμα της εταιρική συμφωνίας σε σχέση με το Μεξικό και συζητήσαμε αυτό. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα φλέγοντα όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ για αυτές τις συμφωνίες. Πολλές άλλες συμφωνίες που συζητήσαμε δεν έχουν αυτό το οικονομικό βάρος και αυτή την οικονομική εμβέλεια και έτσι δεν υπάρχει η αναγκαιότητα να εξεταστούν όλα αυτά με αυτόν τον τρόπο. Επειδή όμως συμβαίνει αυτό τώρα εδώ, με τη ΣΥΠΑ και επειδή οι εναλλακτικέ δυνατότητες ε, ε, για τους εταίρους της Τελωνιακής Ένωσης πρέπει να εξεταστούν, πρέπει να προχωρήσουμε έτσι. Ευχαριστώ. Εσείς παρακαλώ έχετε τον λόγο σώματος των Πρασίνων. Συμφωνώ. Πρέπει πραγματικά αυτό το θέμα να το θέσουμε. Υπάρχει μείζον θέμα, μείζον ζήτημα για την Τουρκία. Επίσης πιστεύω ότι και σε σχέση με άλλες ε, συμφωνίες εμπορίου έχουν τα θέματα των εμπορευμάτων αυτών στις εμπορικές συναλλαγές αλλά δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα, δεν ισχύει η αμοιβαιότητα. Πρέπει λοιπόν να εξεταστεί αυτή η πτυχή. Ευχαριστώ. Εσείς παρακαλώ έχετε τον λόγο από την Ενωτική Αριστερά. Ο κύριος Μέρφυ. Δεν υπάρχει ζήτημα, ότι υπάρχει ζήτημα εδώ για την Τουρκία σίγουρα όμως πρέπει να εξετάσουμε την χρονική αλληλουχία μέσα σε αυτό το πλαίσιο και για την προφορική ερώτηση. Σε σχέση με αυτά τα θέματα, δύο παρατηρήσεις. Η επιδείνωση της κατάστασης στην Τουρκία είναι η πρώτη παρατήρηση. Η σκοτώθηκε ένας διαδηλωτής ε, πριν από μια εβδομάδα περίπου. Ε, τον χτύπησε μια βόμβα δακρυγόνου, δακρυγόνων στο κεφάλι και βλέπουμε την επιθετικότητα της αστυνομίας που ε, παρεμβαίνει ιδιαίτερα επιθετικά. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και το θέμα της Τουρκίας και το γεγονός ότι δεν υλοποιεί τις υποχρεώσεις η Τουρκία εναντί της Κύπρου. Δεν επιτρέπει τα, τα κυπριακά αγαθά να έχουν πρόσβαση σε τουρκικούς λιμένες, ε, λέει ο κύριος Μέρφυ, το ελάχιστο που μπορώ να πω είναι ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην προφορική ερώτηση μία αναφορά στις υποχρεώσεις που απορρέουν για την Τουρκία σε συναφή θέματα όσον αφορά για παράδειγμα την Κύπρο και να μπορέσει η Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτή την πτυχή. Επίσης πρέπει να ε, θέσουμε εδώ τον πύχη υψηλά. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα μπορεί να παρέμβει. Εσείς παρακαλώ έχετε τον λόγο. Thank you, Chairman. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να συνεισφέρουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή τη συζήτηση. Προσβλέπουμε στο να τεθεί η προφορική ερώτηση όταν θα έχει ολοκληρωθεί σε σχέση με τη διατύπωση Συμμεριζόμαστε κάποιες από τις επιφυλάξεις και ανησυχίες που διατυπώθηκαν, για παράδειγμα σε σχέση με την κατάσταση όσον αφορά την Τελωνιακή Ένωση, σε σχέση με τα θέματα ημερήσιας διάταξης από πλευράς ΕΕ. Είναι κάτι που έχει δυσκολίες η Τουρκία, δημιουργούνται δυσκολίες για την Τουρκία σχετικά ακριβώ επειδή κάποιες από τις συμφωνίες ε, ελευθέρου εμπορίου με τους εταίρους μας αρνούν κάποιοι να ε, ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Δεν είναι τόσο πολύ και δεν είναι τόσο σημαντικό το θέμα όσον αφορά τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών ως θέμα αρχής, αλλά δημιουργείται ένα πρόβλημα. Αυτό το θέμα συζητήθηκε με τους Τούρκους εταίρους μας ε, επί αρκετό χρονικό διάστημα. Έχει συνειδητοποιήσει πολύ καλά το τι συμβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να πω ότι υπάρχει μια κοινή συνεννόηση και κατανόηση από αμφότερες τις πλευρές για τη δυσκολία αντιμετώπισης αυτού του θέματος. Και σε σχέση με την τελευταία παρέμβαση που έγινε, ένα από τα θέματα τα οποία τέθησαν επειδή δεν υλοποιεί πλήρως ε, η Τουρκία τις υποχρεώσεις της από την Τελωνιακή Ένωση με όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, βλέπε Κύπρο, αυτό δημιουργεί δυσκολίες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΕ να δείχνει μεγαλύτερη ανταπόκριση προς την Τουρκία. Τούτου λεχθέντος κάνει ό,τι μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναντι της Τουρκίας για να υπάρξει η δυνατότητα διαπραγμάτευσης με τους εταίρους. Όχι μόνο από πλευρά Τη ε, της έναρξης ήδη ή το δυνατόν νωρίτερα με τους ε, ε, διαπραγματευόμενους εταίρους να προχωρήσει το θέμα για τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Επίσης και η ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων με τους Τούρκους εταίρους μας μπορεί να είναι μια δυνατότητα όσον αφορά την ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητήσαμε από τους Τούρκους ε, συναδέλφους να μας αναφέρουν τις δυσκολίες που δημιουργούνται για εκείνους όπως βλέπουν εκείνοι τα πράγματα όταν έρχεται η ώρα διαπραγματεύσεων με τέτοιους εταίρους και όχι μόνο να μας αναφέρουν τις δυσκολίες που βλέπουν αλλά και το ποια είναι τα διαφορετικά αυτά θέματα και τα θέματα τα οποία δημιουργούν τριβές και προβλήματα υποσχεθήκαμε ότι θα τα σημειώναμε και θα τα λαμβάναμε υπόψη ώστε να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε να επιληθούν. Τώρα για τις ε, παρατηρήσεις ε, που έγιναν σε σχέση με αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις προσβλέπουμε στο να δούμε αυτή την ερώτηση και να δούμε ποια αντιμετώπιση θα, ποιας αντιμετώπιση θα τύχει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μετίν Καζάκ για να ολοκληρώσετε. Μου φαίνεται ότι δεν υπάρχει περιθώριο όπως ας το αφήσουμε από την ε, λίστα ψηφοφορίας αύριο. Κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν έχουμε κοινό συμπεφωνημένο κείμενο με τις πολιτικές ομάδες, δεν θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το σχέδιο για την επόμενη ψηφοφορία. Χαίρομαι όμως που υπάρχει κοινή συνεννόηση και πιστεύω ότι αυτό το ζήτημα θα πρέπει να συζητηθεί, να ενημερωθεί η Κομισιόν. Επίση, χαίρομαι που η Κομισιόν δείχνει κατανόηση και βούληση να συζητήσει επί του ζητήματο. Η βασική μα ιδέα είναι ότι θα πρέπει να δούμε συγκεκριμένα ποιες διαδικαστικές πτυχές θα μπορούσαν να ακολουθηθούν ώστε να μπορέσει να εξισορροπηθεί αυτή η ασύμμετρη κατάσταση διότι έγιναν συγκεκριμένες προτάσεις από το τουρκικό Υπουργείο Οικονομίας και εμείς ε, αναμένουμε όχι μόνο σε επίπεδο διοίκησης αλλά και από το υψηλότερο δυνατό επίπεδο της Κομισιόν να λάβει μια απόφαση ακόμη και σε επίπεδο Συμβουλίου ώστε να μπορέσουμε να προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού. Φυσικά πίσω από αυτά βρίσκονται πολλά πολιτικά θέματα. Καλό πιστεύω όμως ότι θα ήταν να εστιαστούμε σε αυτές τις οικονομικές και εμπορικές πτυχές. Θα μας βοηθήσουν ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ψηφοφορία στην Επιτροπή πιθανώς ε, στην επόμενη συνεδρίασή μας τον Οκτώβριο. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό όσον αφορά τη διατύπωση της προφορικής ερώτησης. Αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα, θα πρέπει να συμφωνήσουμε για το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Θα ακολουθεί τώρα η συνεδρίαση συντονιστών. Θα ζητήσω... Δεν παρευρίσκονται ακόμα όλοι εδώ, συνεπώς χρειάζεται να κάνουμε μια, ένα διάλειμμα μέχρι τις 5.30. Εδώ ολοκληρώνεται η δημόσια συνεδρίαση σήμερα. Όσοι λοιπόν δεν μπορούν να μείνουν για τη συνεδρίαση συντονιστών, παρακαλώ να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Ευχαριστώ. Έχουμε ολοκληρωσία σήμερα. Τα λέμε αύριο. Συνεδρία συντονιστών θα ξεκινήσει σε μισή ώρα.